Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας μέρα. Πριν ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, θα ήθελα να καλωσορίσω πρώτα απ' όλα την ομάδα που πρόκειται από την Ακιτέν της SNCF, των Γαλλικών Σιδηροδρόμων. Θα είναι εδώ για λίγο μαζί μας. Καλώ ήρθατε λοιπόν στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού είστε ένας παράγοντας κλειδί. Ε, ξέρετε, για τα αισθήματα των σειρόδρομων, ελπίζω να ξαναέρθετε, διότι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι λυπάμαι που σας ανακοινώνω ότι αξιαγάπητος και μεγάλος Walter Goss 24 ώρες 24 είναι εδώ αυτός ο άνθρωπος έτσι παρακολουθεί ό,τι κάνουμε μου στέλνει και whatsapp για να μου θυμίσει πράγματα που πρέπει να κάνω είναι ο φύλακας άγγελος της Επιτροπής μας Walter μου επιτρέπεις ε, σου μιλήσει στον ελληνικό. Θέλω να σε συγχαρώ για την επαγγελματικότητά σου. 134 συνεδριάσει τη επιτροπή Μεταφορών, 66 συνεδριάσεις συντονισμού, όπου υποφέραμε όλοι μαζί, από το 2012 στο 2019 και πρέπει να σας πω ότι βεβαίως δεν φεύγετε από τον Νίκο μας, θα πάρει στην Επιτροπή Ήτρε. Δεν είναι και άσχημα. Πάντως ε, σας αφήνουμε να φύγετε έτσι με μεγάλη στενοχώρια. Θέλουμε κυρίως να σας ευχαριστήσουμε για να σας πούμε ότι η Επιτροπή Μεταφορών είναι το πρώτο σας σπίτι κατά κάποιο τρόπο και θα σας παρακολουθούμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω στο όνομα της Επιτροπής μας συγχαρητήρια για το έργο σας και στο όνομα των συναδέλφων να σας ε, συγχαρώ. Θέλετε να πείτε κάτι, Βόλτερ, oh. όχι, είστε υπερβολικά συγκινημένος. Και έχουμε βεβαίω και τον αντικαταστάτη, τον κύριο Κλάου Μπάγερ. Έτσι είναι ψηλά ο πύχη, κύριε Μπάγερ. Κλάου. Α, έχετε ήδη εδώ βλέπω κάποιους φαν στην Επιτροπή Μεταφορών, δεν το γνώριζα. Καλώς ήρθατε. Ξέρετε εδώ είναι εξαιρετικά επαγγελματική η προσέγγιση μας. Ορισμένες φορές υπάρχουν εντάσεις, αλλά καταφέρουμε να τα βρούμε. Εσείς πλέον είστε στη θέση του οδηγού. Ο οδηγός βέβαια για μας τους οικολόγους δεν μας αρέσουν τόσο τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα. Καλώς ήρθατε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ξεκινούμε τις εργασίες μας. Η μέση διάταξη μπορεί να εγκριθεί εφόσον δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Θα ήθελα να καλωσορίσω δύο νέα μέλη της γραμματείας της ΤΡΑΝ. Α, όχι, το κάναμε αυτό. Το κάναμε αυτό. Όμως, έχουμε και την κυρία Λογόνς Βατχά. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Έρχεται από τη γραμματεία Ήτρε. Ουσιαστικά εδώ έχουμε μια σκάντζα και θα είναι η βοηθός ε, στην Επιτροπή μας πλέον. Ε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Τραμ. Έχουμε όμως άλλη μια αναχώρηση. Η Βέρα Γεωργίευα, α, ασθενή. Δεν ήθελε να έρθει να τα αποχαιρετήσουμε από τη στενοχώρια της. η οποία ερχόταν στη γραμματεία επίσης ε, εξαιρετικά ευσυνείδητα και αυτή στην Επιτροπή Ήτρε και θα περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να ελέγξω εάν υπάρχει απαρτία πολύ ωραία κύριε Μπαχ Έχετε τις κάρτες σας. Allez, Ψηφίστε ναι, όχι, δοκιμαστικό είναι και αλλιώς, αποχή, ό,τι θέλετε. C'est bon, il n'y a pas de, pas trop de en trop, Εντάξει, δεν περισσεύει κανείς από κανένα, πολιτική ομάδα. Πολύ ωραία. Ξεκινούμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα με τον εισηγητή, τον κύριο Ράντος. Θέλετε το λόγο κύριε Ράντος. Παρακαλώ. Chair, σας ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Πρόεδρε. Πρόκειται εδώ για την ε, συμφωνία με τις ε, Φιλιππίνες. Σύμφωνα με τούτη τη συμφωνία υπάρχει η δυνατότητα να υπήρχε μάλλον πριν η δυνατότητα να, ε, απορρίπτει ή να ανακαλεί ή να αναστέλει άδειε εκμετάλλευση ε, σε αερομεταφορείς ε, οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι σε άλλη χώρα. Είχαμε μετά την απόφαση του δικαστηρίου το οποίο προστατεύει τις αεροπορικές εταιρείες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μετά ξεκίνησε λοιπόν η Κομισιόν διαπραγματεύσει ε, με την Δημοκρατία των Φιλιππίνων. Αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, ολοκληρώθηκαν και τον προηγούμενο Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς δηλαδή υπογράφτηκε η συμφωνία και πλέον ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την συνένεσή του μέσω της ψηφοφορία αυτής στην οποία σα ζητώ η Επιτροπή μα να υπερψηφίσει. Πολύ ωραία. Άρα ψηφίζουμε για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Φιλιππινών όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των αερομεταφορών ε, και αρχή η συνεδρίαση. Η ψηφοφορία, συγγνώμη, ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ω, πάρα πολύ ωραία, ομόφωνα. Εξαιρετική δουλειά που κάνατε. Μπράβο σας και συγχαρητήρια. Ça pour dire c'est du consensus, c'est du consensus. Αυτό κι αν είναι συνένεση. Oh, mais je vous avais pas vu. Comment ça va? Bon. Désormais, on passe au deuxième vote concernant l'objection au règlement délégué. Περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία για την οδηγία 2010-40 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τη χρήση του ETS θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ρικέ. Παρακαλώ. Ε, όσο και αν αγαπώ την Επίτροπό μας και ε, τον εισηγητή και την εισηγήτρια την αγαπητή Γκεζίνε Μάισνερ που υποστηρίζει την πρόταση, εγώ θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο ε, θα πρέπει να προβάλλουμε αντίρρηση. Πράγμα που δεν το συνηθίζω, αλλά τι να κάνουμε. Αρκετοί από εσά ε, το γνωρίζετε γιατί το έχετε υποστεί. Το γεγονός ότι υπήρξε αντίρρηση έχει ανοίξει ε, ένα ολόκληρο κύκλο αντιφατικών ε, πληροφοριών, γιατί πρόκειται για δύο διαφορετικές τεχνολογίες. Η μία βασίζεται στο Wi-Fi και άλλη στην 5G. Ε, ξεκίνησε λοιπόν μια ολόκληρη εκστρατεία πληροφόρησης ε, με δύο στρατόπεδα, ο ένας υπέρ της μίας και ο άλλος υπέρ της άλλης ε, Εγώ δεν θέλω να φέρω αντιμέτωπη μια τεχνολογία απέναντι στην άλλη και τούμπαλη. Δεν είναι αυτή η έννοια της αντίρρησης που σας προτείνω σήμερα να υποστηρίξετε. Ακούσαμε λοιπόν σε αυτή την αντιφατική εκστρατεία πληροφόρησης επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα ως προς το αν είναι διαθέσιμη η τεχνολογία, ε, ποια είναι η βιομηχανική επιλογή, η φύση της, οι επιδόσεις της. Ε, ακούσαμε επιχειρήματα οδικής ασφάλειας, ακούσαμε επιχειρήματα για τις επιδόσεις με τη στενή έννοια ως προς την ε, ασφάλεια και τη μη δυνατότητα παραβίασης και τη γενική στρατηγική της ψηφιακής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Ακούσαμε λοιπόν διάφορα επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα και θα μπορούσε κανείς να πει ότι σχεδόν όλε όλες οι πτυχές φωτίστηκαν και από τις δύο μεριές. Ψηφιακή βιομηχανία, αυτοκίνητο βιομηχανία, για διάφορα άλλα ενεχόμενα μέρη και μεταξύ αυτών και τους χρήστες. Συμπέρασμα, όταν έχουμε μια τέτοια εκστρατεία με διάφορα επιχειρήματα, τα οποία ευσταθούν ε, πολύ ε, εκατέρωθεν, το λιγότερο που μπορεί κανείς να πει είναι ότι υπάρχει αμφιβολία. Αξίζει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτά τα επιχειρήματα Αλλά τώρα επικρατεί και κάποια αγωνία για το τι θα πρέπει να επιλέξουμε και ποιο θα ήταν το σκοπιμότερο. Το θέμα είναι τι προτεραιότητα δίνει κανείς σε ποια επιχειρήματα και ποια προτιμάει. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω διάφορα πράγματα. Πρώτον, αυτή η αμφιβολία είναι ιδιαίτερα έντονη ε, και τη συμμερίζονται πολλοί ε, φορείς, οι περισσότεροι και μάλιστα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, γιατί όπως γνωρίζετε, ο αντιπρόεδρος που είναι αρμόδιος ή αντιπρόεδρος που είναι αρμόδια για τα ψηφιακά ε, ε, έστειλε μια επιστολή που διαφωνεί με αυτή την κατεξουδότηση πράξη. Είναι αρκετά ενοχλητικό αυτό. Δεύτερο, κανείς στον κόσμο δεν έχει επιλέξει τη συγκεκριμένη τεχνολογία είτε έχουν επιλέξει την άλλη, όπως είναι η Κίνα, είτε η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, ε, είτε έχουν σεβαστεί την τεχνολογική ουδετερότητα κάποιες χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα σήμερα στα μεγάλα μπλοκ της παγκοσμιοποίησης κανένα δεν προέβη στη συγκεκριμένη επιλογή. Και το τρίτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι βρισκόμαστε σε περίεργη συγκυρία χρονικά στο τέλος της θητείας με ε, τις συγκεκριμένες συνθήκες ε, παρευρίσκονται εδώ 31 βουλευτές οι περισσότεροι είναι αναπληρωτές και τους ευχαριστώ αλλά δεν είμαστε τώρα σε μια έτσι πάρα πολύ ήρεμη περίοδο και γαλήνια και ένα τελευταίο αν κάνουμε αυτή την επιλογή, είμαστε απολύτω αντίθετοι προ την τεχνολογική ουδετερότητα που πάντα προκρίναμε σε όλε τι επιλογέ μα. Συμπέρασμα. Πιθανότατα, χωρί να θέλω να προεξοφλήσω τίποτα ή να προωθήσω καμιά τεχνολογία απέναντι στην άλλη, θεωρώ ότι οι αμφιβολίες είναι περισσότερο από ε, σοβαρές και τα επιχειρήματά τους και στη συνέχεια δεν υπάρχουν τίποτα ακράδαντα επιχειρήματα για να πούμε ότι είναι τόσο επίγοντο το θέμα ώστε να αποφασιστεί ε, τέτοιες ώρες και σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε και την ε, αναταραχή. Άρα, νομίζω ότι είναι λογικό να εκφράσουμε κάποιες αμφιβολίες και να φανούμε προσεκτικοί και συνεπτοί γιατί αυτή η επιλογή ό,τι και αν διαλέξουμε είναι σημαντική και μας δεσμεύει πάρα πολύ προς τη μία κατεύθυνση ή την άλλη ε, για τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να μείνουμε εκεί. Εγώ με την αντίρρηση αυτή λοιπόν δεν σας ζητώ να υποστηρίξετε μια τεχνολογία απέναντι στην άλλη, σας ζητώ να εκφράσετε την αμφιβολία σας γιατί τίθενται πολλά ε, ερωτηματικά, αναπάντητα ερωτήματα. Κανείς δεν έχει επιλέξει σήμερα από τους φορείς παγκοσμιοποίηση τη συγκεκριμένη οδό, το αντίθετο μάλιστα. 15 μέρες έχει που ήρθε η τεχνολογία 5G και στη Γερμανία απέριψαν ε, την τεχνολογία Wi-Fi στη βιομηχανία και επιλέγουν το 5G. Λοιπόν, υπάρχει λόγος να αφιβάλλει κανείς και να επιδείξει ψήνεση και επιφυλακτικότητα. Θα πρέπει να γίνει αυτή η επιλογή, δεν λέω, αλλά όχι τώρα, γιατί μας δεσμεύει πάρα πολύ και εμάς και το ψηφιακό μας μέλλον και τη βιομηχανία και μάλιστα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα και αποκρισταλώσει άποψη. Γι' αυτό κυρία Πρόεδρε, ε, ας είμαστε προσεκτικοί να το ξανασκεφτούμε με την ησυχία μας και να μην μπούμε βεβαιασμένα σε μια επιλογή που δεν είναι ε, προφανώς μη αναστρέψιμη, αλλά θα μας δεσμεύσει για τα επόμενα χρόνια σε μια αμφίβολη, ε, δεν είπα αμφιβλεγόμενη, ε, επιλογή. Χρειάζομαι 7 συναδέλφους για να κάνουμε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση γιατί πραγματικά θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό και να τοποθετηθούμε γιατί θα το ξαναβούμε μπροστά μας του επόμενου μήνες και χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρικέ. Για να γίνει κατανοητό σε όλους, ο εισηγητής της αντίρρησης ο κύριος, ε, είναι ο κύριος Ρικέ, αλλά η εισηγήτρια είναι η κυρία Μάισνερ όσον αφορά την κατεξουσιοδότηση της πράξης. Κυρία Μάισνερ, θέλετε να πάρετε το λόγο, φαντάζομαι ναι. Ναι, εντάξει είναι απολύτω θεμητό να προβάλλει κανεί αντίρρηση σε μια τέτοια κατεξοδότηση πράξη. Το είπε Ντομινίκ Ρικέ, ε, αλλά δεν είπε κάτι άλλο. Ε, ότι συνήθω έχουμε ένα τρίμηνο για να αποφανθούμε αν είμαστε υπέρ ή κατά. Τώρα είναι δίμηνο αυτή η περίοδο. Βέβαια, καλύτερο θα ήταν να έρθει νωρίτερα η πρόταση για να προλαβαίνουμε, αλλά τι να κάνουμε δεν είχε προκύψει ακόμα. Αυτά για τα χρονικά. Αλλά αν κανεί είναι απόλυτα πεπισμένος ότι μπορεί να πάρει μια απόφαση και είναι σωστή, γιατί να μην την λαμβάνει. Δεν έχουμε εξαντλήσει πάντα το τρίμηνο, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά είπε, Ντομινίκ, ότι ο Επίτροπος Άνσιπ ε, είχε κάποιε επιφυλάξει στην αρχή, μάλιστα και έστειλε και επιστολή. De facto όμως, αφού... Ε, το συζήτησε μαζί του η Βιολέτα Μπόλτς και οι άλλοι αρμόδιοι επίτροποι, του είπα να το φέρει στο κολέγιο και τότε έκανε πίσω και είπε, α ναι, το ξέρω ότι οι περισσότεροι επίτροποι θεωρούν ότι αυτό που προτείνεται είναι εντάξει. Αλλά ο ίδιος είχε τις επιφυλάξεις του, τις οποίες απέσυρε. Αυτά λοιπόν είναι παροχημένα πλέον πράγματα και η πλειοψηφία, η πλειονότητα των επιτρόπων προχώρησε προς τα εκεί. Η τεχνολογική ουδετερότητα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεχνολογία η οποία είναι έτοιμη, είναι το 5G, ε, ε, ε, μάλλον όχι το 5G, είναι το Wi-Fi και προβλέπεται κιόλας εκ των υστέρων ε, να γίνουν συμβατές οι δύο τεχνολογίες. Υπάρχει κάποια χρονική στέρηση ακόμα, αλλά εγώ το συζήτησα με διάφορες εταιρείες που μου είπαν ε, ότι όταν οριμάσει και άλλη τεχνολογία μπορεί να συνδυαστεί με την πρώτη. Ε, αν ξεκινήσουμε τώρα το G5 μπορούμε να προχωρήσουμε για την ε, επικοινωνία μεταξύ των ε, οχημάτων, car to car λέγεται αυτό, ε, για να συνεισφέρουμε και για την οδική ασφάλεια. Γιατί οτιδήποτε μπορεί να αποφύγει τα τροχαία και τα δυστυχήματα ήταν προτεραιότητά μας. Εγώ τα μελέτησα αυτά τα θέματα όλα από την αρχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας στηρούσε συνέχεια ενημερούς για τις καινοτομίε, για, τα νέα δεδομένα, τις εξελίξεις κτλ. Και, τα λοιπά, και τις τελευταίες τεχνολογίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την εντολή αυτή και με διάφορες εκθέσεις και με την νομοθεσία να μας παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και να προσαρμόζει και τις υποδομές της. Και το κάνει κιόλας. Άρα, εδώ υπάρχουν κάποια εθνικά συμφέροντα τα οποία είναι αντιφατικά και μπορώ να σας τα πω. Υπάρχουν αυτοκινητοβιομηχανίες και στη Γερμανία που λένε ότι περιμένετε γιατί έχουμε ποντάρει στο 5G, αλλά λένε πάμε γιατί είμαστε έτοιμοι οι περισσότεροι θεωρούν ότι θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα αυτό. Ε, είναι λογικό για να είμαστε και, και μπροστά στις παγκόσμιες εξελίξεις και εγώ το ίδιο πιστεύω. Το κοίταξα προσεκτικά. Ξέρω ότι υπάρχουν αφιβολίες, Ευρωπαϊκή Κατά την άποψή μου, αυτό όμω που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι και σωστό και προϊόν ορίμου σκέψεως. Μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε με το G5 και όταν οριμάσει και το 5G, τότε μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Αν προβάλλουμε την αντίρρηση και το φρενάρουμε, φυσικά γίνεται και είναι και δημοκρατικά δυνατό, αλλά χαιρετίσματα. Θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα χρόνο για να αρχίσουμε να δημιουργούμε νέε υποδομέ και θα είναι ένα χρόνο χαμένο. Και πού είναι η οδική ασφάλεια. Το θεωρώ και ανεύθυνο. Και κατά την άποψή μου, αγαπητέ Ντομινίκ, θα πρέπει να απορρίψουμε την αντίρρηση αυτή είπε ότι δεν έχει προτίμηση για καμία τεχνολογία. Συνδυάζονται αυτέ οι δύο τεχνολογίε στο μέλλον στου αυτοκινητοδρόμου. Α αρχίσουμε με τη μία που είναι τώρα έτοιμη και βλέπουμε με την άλλη. Γι' αυτό ζητώ να απορριφθεί αντίρρηση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάισνερ. Λοιπόν, ο κύριος Ρικέ μας ε, ζήτησε ονομαστική κλίση, ψηφοφορία δηλαδή διανομαστικής κλίσης, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν όχι 7 αλλά 10 ε, βουλευτές υπέρ. Ε, ποιοι λοιπόν θα ήταν υπέρ μιας ψηφοφορίας διανομαστικής κλίσεως. Συμφωνείτε να γίνει roll call vote για το κείμενο αυτό. Ψήφισαν όλοι. Ωραία, πέρας έχετε πάνω από 10. Επομένως, ναι, θα έχουμε ψηφοφορία διονομαστικής ω επί του κειμένου σας, κύριε Ρίκε. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. J'ai un petit doute. Bon, allez, allez, je ferme le vote. Pardon. Πέρας. Et c'est adopté. Ken Grinete. Donc, les conséquences... Αυτό σημαίνει αυτό σημαίνει ότι θα συγγράψουμε την αντίρρησή μας, την οποία θα αποστείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα τη στείλουμε στην Ολομέλεια, διορθώνει η Πρόεδρος, και θα εγγραφεί στην Ολομέλεια. Θα έχουμε λοιπόν πάλι το κείμενο αυτό στην Ολομέλεια αυτή τη φορά. Η αντίρρηση πρέπει να περάσει και από την Ολομέλεια. Δεν τελειώσαμε ακόμα, μη φεύγετε, καθίστε. Non, ce n'est pas notre όχι, δεν είναι η τελευταία μας συνεδρίαση. Η επόμενη λοιπόν συνεδρίασή μας θα λάβει η χώρα την 11η Απριλίου. Προσέξτε να είστε όλοι εκεί. Τώρα τελείωσε η συνεδρίαση. Χαίρετε.